So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ladies and gentlemen, colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Καθίστε αν θέλετε. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Η σημερινή συνεδρία μπορεί να ξεκινήσει. Και συνεχίζω στα γερμανικά. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις, προτείνω την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Κυρία Σόιντροβα, ζητάει το λόγο για την ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να παρακαλέσω να αναβληθεί η ψηφοφορία για τις δύο θέσεις αντιπροέδρων, καθώς δυστυχώς δεν είμαστε βέβαιοι πως ο υποψήφιος που θέλουμε να προτείνουμε θα εκλεγεί. Με λύπη μου λοιπόν λέω πως ασκούνται κάποιες πιέσεις. Γι' αυτό θα θέλαμε να μας δοθεί περισσότερο χρονικό περιθώριο για να προχωρήσουμε στις συνομιλίες και διαπραγματεύσεις. Γιατί θέλουμε να υποστηρίξουμε την υποψηφιά μας. Γι' αυτό σας παρακαλώ να αναβληθεί για το Σεπτέμβριο η ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Καμερέβερτ, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Λυπούμε κι εγώ, αλλά δεν συμφωνούμε για την αναβολή σήμερα. Δεν βλέπω τι θα μπορούσε να αλλάξει μέχρι το Σεπτέμβριο. Γι' αυτό παρακαλώ να γίνει σήμερα η ψηφοφορία όπως έχει προβλεφθεί. κυρία Σόιντροβα. Πρόεδρε, αν δεν υπάρχει συμφωνία για την αναβολή, προτείνω την ε, υποψήφια για τη θέση της Ετάρτης ε, Αντιπροέδρου. Επιμένω όμως για την αναβολή. Μάλιστα, έχω δύο προτάσει. Η μία αφορά αναβολή και των δύο ψηφοφοριών για το Σεπτέμβριο. Ψηφίζουμε αυτό πρώτο, που είναι η πιο ε, ριζική πρόταση. Η δε άλλη αφορά την αναβολή για την ψηφοφορία τη τέταρτη, αντιπρόεδρου. Θα ψηφιστεί το έτοιμο αυτό στη συνέχεια. Αλλά θέλω να επισημάνω ότι Έχουμε ορισμένους αναπληρωτές σήμερα εδώ και γι' αυτό θα ήθελα, εάν τυχόν και δεν έχουν δηλωθεί όλοι οι αναπληρωτές, εάν δεν έχουμε δει ο κύριος Ζαγοράκης αντικαθίσταται τον κύριο Βίνκλερ, για τους σοσιαλιστές δημοκράτες ο κύριος Δεμπλάνκο, από το Renew Europe η κυρία Μέλτσιορ, αντικαθίσταται τον κύριο από την κυρία Μούλτινγκ, κύριος Μπουτκό. Αντικαθιστά τον κύριο Κάνκο, την κυρία Κάνκο, στο συγγνώμη. ECR. Κατερίν Κριζέ, Ντόμινικ Μπίλτ. Και μετά για την κυρία Φόξ, η κυρία Τζέμα. Έχουμε αρκετές αναπληρώσεις σήμερα βουλευτών λόγω των εκλογών. Παρακαλώ. To press, to press the button to activate. This one? Yes. Uh, Anne-Sophie Pelletier for... Γεωργιούλης. Γεωργιούλης. Anne-Sophie Pelletier, αντικαθιστά τον κύριο Γεωργούλη. Für die Mitteilung Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Άλλος ε, που αντικαθιστά. Όχι. Ερωτώ λοιπόν, έχετε όλοι τις κάρτες σας για την ψηφοφορία. Είμαστε εντάξει. Δεν σας άκουσα. Äh, Μπορείτε να ζητήσετε από τους βοηθούς σας να τρέξουν να φέρουν τις κάρτες για να είμαστε έτοιμοι. Ούτως ή άλλως δεν θα είναι μυστική ψηφοφορία, θα γίνει διανατάσσεως της χειρός. Επομένω, ε, ένα μικρό διάστημα το έχετε το περιθώριο αυτό δηλαδή για να πάνε βοηθοί να φέρουν τις κάρτες. Ωραία, ψηφίζουμε λοιπόν το πρώτο αίτημα για την εκλογή τρίτου και τέταρτου ή τρίτης και τέταρτης αντιπροέδρου. Αναβολή για το Σεπτέμβριο, προκειμένου να εξασφαλιστεί και για τις δύο αυτές θέσεις μια συμφωνία. Ποιος είναι υπέρ της αναβολής? Oui, euh, pour ma part, je pense aussi Πιστεύω και εγώ ότι καθυστερούμε πολύ στο θέμα της αναβολής. Η ομάδα μου λοιπόν είναι κατά της αναβολής σήμερα. Εκτός και αν το ΕΛΚ έχει να προτείνει άλλον υποψήφιο. Ναι, μα ακριβώς αυτό χρειάζεται χρόνο γιατί έχουμε το σύστημα DONT και δεν είναι δυνατόν δυνάμει του συστήματο αυτού να βγει κάποιο να πει τώρα προτείνω άλλον υποψήφιο. Δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη αυτό. Υπάρχουν και άλλε συνομιλίε του ή άλλο αν εξελίξει. Γι' αυτό προτείνω να διατηρηθεί το σύστημα, να τηρηθεί το σύστημα DONT και να δούμε αυτό το, αυτούς τους υποψηφίους. Κυρία Σόεντροβα, στα γαλλικά, ναι. Αντιλα βάνομαι ότι σας προβληματίζει αυτή η κατάσταση. Δεν με ικανοποιεί η ιδέα της αναβολής, αλλά να εξηγήσω γιατί είμαστε βέβαιοι ότι ο κύριος Ανδρέα Μπόσκορς ή η κυρία Μπόσκορς ε, θα είναι πράγματι κατάλληλη υποψήφια, γιατί είναι ένας άνθρωπος πολύ εργατικός και δραστηρίος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αποκλειστεί η δική μας υποψήφια. Πέντε χρόνια τη γνωρίζουμε, έχουμε συνεργαστεί μαζί της και αισθανόμαστε πολύ μεγάλη δυσφορία για την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Ναι, βεβαίως θα ψηφίσουμε. Αλλά αυτό είναι ο λόγος. Και βεβαίως θα συνεχίσουμε με συνομιλίες και διαπραγματεύσεις. Η Πρόεδρος, το πρόβλημα είναι ότι δεν μας επιτρέπει η μυρίσια διάταξη να κάνουμε συζήτηση επί της ουσίας. Γι' αυτό θα ήθελα να γίνει ψηφοφορία αμέσω. Ναι, δεν θα αφήσω δηλαδή να γίνουν άλλες συζητήσεις. Επί της ε, ουσίας ή ε, επί προσωπικών ε, κρίσεων δεν έχουμε περιθώριο να συζητήσουμε τώρα και αυτό ας ψηφίσουμε. Ποιος είναι υπέρ της αναβολής και των δύο ψηφοφοριών, τρίτης και τέταρτης αντιπροέδρου, για το Σεπτέμβριο. Κατά. 14 υπέρ, 14 κατά. Και άρα απερίφθη το αίτημα για αναβολή. Δεύτερο αίτημα. Αναβολή μόνο για την τέταρτη ή τον τέταρτο αντιπρόεδρο. Όχι, να επαληθεύσουμε, εντάξει. Επαληθεύουμε το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας, αλλά δεν έχουν όλες τις κάρτες τους μαζί. Εφόσον δεν είναι και μυστική ψηφοφορία, μπορούμε να μετρήσουμε την ψήφο του κυρίου Αντέμοφ. <laughs> και εγώ δεν έχω τη δικιά μου, την έχασα, αλλά πρέπει να ψηφίσουμε και οι δύο. Κανονικά την έχω κρεμασμένη στην αρμαθιά, αλλά δεν τη βλέπω τώρα. Μπορεί να πέσαμε στην τσάντα μου. Αλλά μπορούμε με την επαληθεύση να το δούμε αυτό. Επαληθεύουμε λοιπόν για την αναβολή, υπέρ της αναβολής παρακαλώ να ψηφίσετε ναι. Επαληθεύουμε. It's not working or? Δεν λειτουργεί. has won too much. Μάλιστα, οι σοσιαλιστές έχουν έναν υπεράριθμο. Να επαληθεύσουμε για άλλη μια φορά ότι δεν έχουν υπεράριθμους ε, οι ομάδε σε σχέση με, το, με τη δύναμή του. So, ich schließe hier mit die το της 13 υπέρ, οι δύο ψήφοι δικέ μας. 15 υπέρ, 15 κατά. Ξεκολουθούμε να έχουμε πατ και άρα απεριφθεί η πρόταση. Και τώρα ψηφίζουμε ε, το δεύτερο αίτημα για αναβολή της ψηφοφορίας για τέταρτο ή τέταρτη αντιπρόεδρο το Σεπτέμβριο. Υπέρ παρακαλώ. Πάλι με ανάταση. Υπέρ. Κατά. Υπέρ. Λοιπόν αποφασίστηκε και έτσι γίνεται σήμερα η ψηφοφορία για τον Ιτρίν τρίτη αντιπρόεδρο και αναβάλλεται η ψηφοφορία για τον τέταρτο. Και περνούμε στις ανακοινώσεις της Προέδρου. Σήμερα λοιπόν διερμηνία ε, έχουμε στις εξής ε, γλώσσες γαλλικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, τσεχικά, ουγγαρικά, λατινικά, πολωνικά, σλοβενικά, βουλγαρικά, σλοβακικά και κροατικά. Άρα δηλαδή έχουμε σχεδόν πλήρη σύστημα, πλήρη κάλυψη των γλωσσών που, στις οποίες προσφέρονται διερμηνία και η Πρόεδρος ευχαριστεί τους διερμηνείς για τη δουλειά του. Ήθελα λοιπόν να σας υπενθυμίσω ότι η συνάντησή μας ε, μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου και επίσης θα ήθελα να ανακοινώσω ότι οι των συντονιστών της 15 Ιουλίου 2019 οι οποίες σας εστάλησαν στις 16 Ιουλίου με ηλεκτρονικό μήνυμα οι ε, αποφάσεις αυτές ε, αν δεν αμφισβητηθούν μέχρι τις 18 Ιουλίου θα θεωρούν εγκεκριμένες. Πάμε στο σημείο υπερτιμών 3 της ε, ημερήσιας διάταξης. Εκλογή του ή της ε, τρίτου ε, αναπληρωτή προέδρου, αντιπροέδρου μάλλον. Πάμε τώρα ε, στα ονόματα. Βίνκλερ, Καρθία Ντεμπλάνκο, Κάριν Μέλχο, Κάνκο, Μπίλντε, Τζέμα, και κύριε Μπετιέ. Αυτά τα ονόματα μου έχουν προταθεί. Ε, αυτοί είναι οι αντιπρόεδροι που θα συμμετάσχουν σήμερα στην εκλογή. Από ό,τι βλέπω αυτοί είναι, δεν προστίθεται κανένα άλλο. Ω εκ τούτου διαπιστώνω ότι έχουμε απαρτία εφόσον έχουμε παρόντα οκτώ μέλη και σήμερα βλέπω ότι είναι παρόντα πολύ περισσότερα από οκτώ μέλη. Θα ήθελα λοιπόν να επισημάνω στην ομάδα ότι εάν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας προκύψει κάποια εκλογή σχετικά με τους πρόεδρους, θα πρέπει να το ανακοινώσετε στην πρόεδρο. Και τώρα ε, θα ήθελα να ακούσω ποιος προτείνεται για τρίτος αντιπρόεδρος. Εμείς ε, για τη, εκ μέρους των σοσιαλιστών προτείνουμε την κυρία Τζούλι Ward. Και ερωτώ, υπάρχουν άλλοι υποψήφοι από ό,τι βλέπω. Όχι, ως εκ τούτου διαπιστώνω ότι η κυρία Τζούλι Ward που είναι πλήρες μέλος ε, της Επιτροπής Πολιτισμού, προτάθηκε από μια πολιτική ομάδα. Η δήλωσή της ε, για τα οικονομικά συμφέροντα και η δήλωση σχετικά με τον κώδικα δεοντολογίας έχει συμπληρωθεί. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την υποψήφια ε, κατά πόσον δέχεται αυτή την πρόταση. Ναι, το δέχομαι φυσικά γιατί είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μένα το ότι μπορώ ε, να αναλάβω αυτό το καθήκον. Έχω την εμπιστοσύνη πολλών ανθρώπων. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ και όσοι με γνωρίζουν από την προηγούμενη θητεία θα ήθελα να ευχαριστήσω κυρίως αυτούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος και θέλω τώρα να ρωτήσω μήπως θέλει κάποιος να προτείνει να υπάρξει μυστική ψηφοφορία. Η κυρία Ζόρντοβα. Θα ήθελα πράγματι να υπάρξει μυστική ψηφοφορία, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά με μυστική ψηφοφορία. Βεβαίως αυτό θα πρέπει να ε, στηριχτεί ε, από τουλάχιστον πέντε. Βέβαια ε, την πρόταση της κ. Ζόντροβα την έχουν στηρίξει οκτώ από την πολιτική της ομάδα που είναι και παρόντες. Ως εκ τούτου η ψηφοφορία θα γίνει μυστική. Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι ε, πράγματι θα γίνει αυτή η μυστική ψηφοφορία γιατί το ζήτησαν τουλάχιστον πέντε πλήρη μέλη της Επιτροπής και θέλω να υπογραμμίσω ότι κάθε μέλος ε, έχει μία ψήφο και έχουμε ΕΛΚ 8, Σοσιαλδημοκράτες 6, Renew Europe 4, Πράσινη 3, η ID 3, ε, το ECR 3, η GUE 2 και οι μη εγγεγραμμένοι δύο ψήφους. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι η ψηφοφορία θα πρέπει κάθε φορά, σε κάθε γύρο ψηφοφορίας, να γίνεται με πλήρη, με απόλυτη πλειοψηφία. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να ε, ψηφίσουμε για την κυρία Τζούλι Γουόρτ, για την τρίτη αντιπρόεδρο. Παρακαλώ ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε με μυστική ψηφοφορία. Μισό λεπτό. Ε, κοιτάξτε, τα κουμπιά, δέστε μπροστά σας. Ε, βλέπετε λοιπόν μπροστά σας. Όπα. Κάτι δεν πάει καλά σήμερα, λέει η πρόεδρος. Κάτι, κάτι δεν πάει καλά. Πολύ δραματικά όλα αυτά. Λοιπόν, έχετε μπροστά μία οπή. Εκεί μπαίνει η κάρτα. Όποιος δεν το γνωρίζει, ε, αν είναι νέο μέλος, ε, θα βάλτε την κάρτα και θα ανάψει το όνομά σας. Αν δεν δείτε το όνομά σας, δεν έχει μπει καλά η κάρτα. Και γι' αυτό σας παρακαλώ να το ελέγξετε όλοι. Βάζετε σωστά την κάρτα. Και μετά δεξιά ε, βλέπετε τρία κουμπιά. Ε, το αριστερό είναι πράσινο, είναι το ναι. Στη μέση το λευκό είναι αποχή και το δεξιά ε, είναι για όχι. Το κόκκινο δεξιά. Λοιπόν, δοκιμή. Τώρα θα κάνουμε μια δοκιμή γιατί σε αυτή την επιτροπή δεν έχουμε ψηφίσει ακόμα με μυστική ψηφοφορία. Και τώρα, ε, εγώ, Ποιος θέλει τον πρόεδρο Πλάσιντο Ντομίνγκο, έτσι για να λέμε. Ψηφίζουμε λοιπόν. Πλάσιντο Ντομίνγκο, πρόεδρος. Ψηφίζετε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ε, ψηφοφορίας. Στην περίπτωση αυτή ψήφισαν 23, 6 αποχές, 5 όχι και 18 ναι. Ως εκ τούτου, θεωρητικά, ο κύριος Πλάσο Ντομίνγκο θα ήταν, θα είναι πρόεδρό μα. Επειδή όμω σήμερα δεν ψηφίζουμε για τον κύριο Ντομίνγκο, αλλά για την Julie ξανά ξαναψηφίζουμε τώρα για την Τζούλι Ward. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Αρχίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορία ψήφισαν ναι και όχι οι 24. Οι 18 υπερψήφισαν ναι δηλαδή, 5 αποχές και 6 καταψήφισαν, 6 όχι. Ως εκ τούτου η κυρία Τζούλι Γουόρτ εξελέγει. Τζούλι, δέχεσαι το αποτέλεσμα της ε, ψηφοφορίας. Τζούλι, δέχεσαι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Ε, υποθέτω ότι εφόσον δέχεται τα συγχαρητήρια, δέχεται και το αποτέλεσμα της ε, εκλογής. Συγγνώμη, ήμουν αποσχολημένη με τα συγχαρητήρια. Προφανώς και δέχομαι την εκλογή. Ε, παρακαλώ, αν έχετε να έρθετε μπροστά στο βήμα, να κάτσετε στη θέση σας. Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπου πρόκειται για τον τέταρτο αντιπρόεδρο, εκλογή τετάρτου αντιπρόεδρου, το αναβάλαμε για το Σεπτέμβρη. Ω εκ τούτου ξεκινάμε τώρα με τις υπόλοιπε ψηφοφορίες. Έχουμε διάφορες ε, ψηφοφορίες. Σήμερα ψηφίζουμε για τρεις ε, εντολές ε, έτσι ώστε να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα Erasmus Plus, για το Greater Europe και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης. Όπως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τα τρία προγράμματα σας έχει παρουσιάσει την άποψή του σε πρώτη ανάγνωση. Η Φιλανδική Προεδρία είπε ότι είναι πρόθυμη τις διαπραγματεύσεις να τις ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν και επειδή είναι προς όφελός μας να μην καθυστερήσει η ψηφοφορία, γι' αυτό θα πρέπει να προλιάνουμε το έδαφος, να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Και αυτό θεωρώ ότι είναι σωστό, γιατί το 2021 θα έχουμε ένα νέο πρόγραμμα και μέχρι το 2020 δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε την παράκληση να συμφωνήσετε έτσι ώστε να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατόν τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο έτσι ώστε το πρόγραμμα να καταστεί δυνατόν να ολοκληρωθεί και από το 2021 να μπορούμε πλέον ε, να ε, συνεχίσουμε την εφαρμογή των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελος των νέων και των δημιουργών. Επιτρέψτε μου να επισημάνω και ορισμένα άλλα πράγματα. Άρθρο 72 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρει ότι το Κοινοβούλιο εφόσον έχει δεχτεί σε πρώτη ανάγνωση το αποτέλεσμα, τότε προκύπτει εντολή και η αρμόδια επιτροπή μπορεί ανα πάσα ώρα και στιγμή ε, αργότερα με πλειοψηφία των μελών να αποφανθεί επί της έναρξης των δύο Άρα δηλαδή 16 ναι για κάθε μία από τις τρεις εντολές και γι' αυτό προτείνω να ξεκινήσουμε ευθύ αμέσω με τις ε, ψηφοφορίες. Ή μήπω θέλει σε σημείο αυτό κάποιο από τους συζητητές να λάβει το λόγο. Από ό,τι βλέπω όχι, Ω εκ τούτου μπορούμε να προχωρήσουμε στις ε, ψηφοφορίες. Ψηφίζουμε καταρχήν για το πρόγραμμα Erasmus+. Ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά και ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. 27 ναι, μία εποχή, ε, μία ψήφος ε, κατά. Ως εκ τούτου, μόλις είναι έτοιμο το Συμβούλιο, μπορούμε να ξεκινήσουμε τις ε, διαπραγματεύσεις. Πάμε τώρα στη δεύτερη ψηφοφορία. Πρόκειται για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα Creative Europe. Ψηφίζουμε, παρακαλώ. Άρχεται η ψηφορία. Ψηφίζουμε, παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Και εδώ 27 ναι, μία αποχή και μία ψήφος κατά. Ως εκ τούτου έγινε δεκτή ε, δεκτό το αίτημα. Πάμε στο, στην επόμενη ψηφορία. Πρόκειται για την ψηφορία σχετικά με την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων ε, πάντα σε σχέση με το πρόγραμμα για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Πέρα της ε, ψηφοφορίας 23 ναι, 2 αποχές και 3 όχι. Και εδώ λοιπόν με μεγάλη πλειοψηφία ε, ψηφίσαμε υπέρ της ε, έναρξης των διοργανικών διαπραγματεύσεων. Και πάμε τώρα στο σημείο υπερθμών 8 της ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για το σχέδιο προπολογισμού του 2020, πρόκειται για την παρουσίαση των τροπολογιών στο ε, σχέδιο προπολογισμού από την άποψη και από το πρίσμα του συντάκτη της γνωμοδότησης. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η Κομισιόν στις 5 Ιουνίου του 2019 δημοσίευσε το σχέδιο του προπολογισμού πολισμού για το έτος 2020. Όλα τα σχετικά έγγραφα, ε, τα έγγραφα αυτά στάλησαν στα μέλη της Επιτροπής στο πλαίσιο της διαδικασίας. Υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα είναι η τοποθέτηση της Επιτροπής μας για το σχέδιο προπλογισμού, η θέση μας η οποία θα παρουσιαστεί στις 4 Σεπτεμβρίου και το δεύτερο είναι οι τροπολογίες που αφορούν το ίδιο το σχέδιο του προπολογισμού και επί των οποίων θα ψηφιστεί ήδη στις 4 Σεπτεμβρίου. Η κυρία Κάμερεβερτ, η συγγήτρια, σήμερα θα μας παρουσιάσει τι είδους τροπολογίες προτίθεται να υποβάλει για το σχέδιο προπλογισμού. Και πριν σου δώσω το λόγο, Πέτρα, θα ήθελα να επενθυμίσω ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών ε, τελειώνει στις 25 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα. Οι τροπολογίες με βάση την απόφαση των συντονιστών 15 Ιουλίου πρέπει να κατατεθούν στην αγγλική γλώσσα και όλες οι προτάσεις για πιλωτικά προγράμματα ή προκατακτικά μέτρα θα πρέπει να κατατεθούν εκ νέου. Και αυτό οφείλεται στο ότι πρέπει να τηρήσουμε κάποιες προθεσμίες. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και αυτό οφείλεται στο ότι ε, θέλαμε βέβαια να δώσουμε τη δυνατότητα και στα νέα μέλη να καταθέσουν νέε τροπολογίε. Γιατί αν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία όπω προβλεπόταν πριν από τι εκλογέ, δεν θα είχαν την ευκαιρία αυτή τα νέα μέλη. Κατ' εξαίρεση λοιπόν, σα παρακαλώ να δεχτείτε αυτή την προπόθεση, αυτόν τον περιορισμό και Πέτρα έχει το λόγο για 15 περίπου λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ αγαπητή Σαμπίνα, αγαπητοί συνάδελφοι. Ξεκινήσαμε ήδη την Άνοιξη του 19 τη διαδικασία για τον προϋπολογισμό. Τον Απρίλιο μάλιστα η Επιτροπή μας απέστειλε και επιστολή στην ε, Επιτροπή προϋπολογισμών επισημένοντας ε, για τον δημοσιονομικό σχεδιασμό από το 2020 τις προτεραιότητές μας. Είδα αυτή την εβδομάδα τους συντονιστές ε, για να συζητήσουμε. Μάλλον ορίσαμε αυτή τη βδομάδα τους συντονιστές. Ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε. Με ενδιαφέρει βέβαια να καταθέσουμε αυτή την ε, τροποποίηση στον κανονισμό και να ακούσω και να λάβω υπόψη για τις δικές σας τις τροπολογίες μέσα στο κείμενο. Το πολιτικό κείμενο της γνωμοδότησής μας δηλαδή. Οι προτάσεις δικές μας για τον προϋπολογισμό θα πρέπει να εστιάζονται σε τρία σημεία. Πρώτον στις προτεραιότητες της Επιτροπής μας που αναφέρονται άλλωστε και στην επιστολή που αποστήλαμε στην Επιτροπή των Προϋπολογισμών ειδικότερα την διαφύλαξη του επίπεδου χρηματοδότησης για το Erasmus Δημιουργική Ευρώπη και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, αλλά και για το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες. Και επίσης θέλουμε να εξετάσουμε ποια είναι η θέση του Συμβουλίου όπως ορίστηκε τον Ιούλιο του 2019 και σε σχέση με τα πιλωτικά προγράμματα και τα μέτρα που θα τα αφορούν. Προτείνω λοιπόν, όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο στον προϋπολογισμό σε σχέση με αυτά που προτείνει η Επιτροπή, που ελπίζω ότι θα μπορέσει να γίνει δεκτό και από το Συμβούλιο για τα προγράμματα στα οποία έχουμε αρμοδιότητα και στα οποία φαίνεται σημαντική πρόθεση περικοπών ε, γενικά, ενώ για το Erasmus ε, Plus ε, δεν υπάρχουν περικοπές, αλλά δεν μπορούμε να δεχθούμε για τα υπόλοιπα προγράμματα στα οποία έχουμε αρμοδιότητα θα επιβάλλει το Συμβούλιο σημαντικές περικοπές. Το Erasmus Plus, το Creative Europe, το Σώμα εθελοντών αλλά και το πρόγραμμα για τους πολίτες της Ευρώπης ξέρουμε ότι έχουν τεράστια συμβολή στην ε, ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πολίτες. Δεν έχουμε παραλείψει καμία ευκαιρία και εμείς και η Επιτροπή να υπογραμμίσουμε πόσο σημαντικό είναι ε, το ζήτημα αυτών των προγραμμάτων και η χρηματοδότησή τους, αλλά φαίνεται ότι πως ε, το Συμβούλιο κοφεύει. Οι περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο είναι απολύτως απαραδεκτές για μένα δεν χρειαζόμαστε λιγότερα, αλλά περισσότερα κονδύλια για τα προγράμματα αυτά, για το Δημιουργική Ευρώπη, για το πρόγραμμα για τους πολίτες που έχουν χρόνια υποχρηματοδότηση, άλλωστε και εμείς, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ίδια έχει μιλήσει και για ποσοστά απόρριψης 70%, όχι γιατί ήταν κακά τα προγράμματα τα οποία ε, είχαν κατατεθεί, αλλά γιατί δεν υπήρχαν τα κονδύλια για να τα καλύψουν. Και έτσι προτείνω για το Erasmus για το Δημιουργική Ευρώπη, αλλά και για το Ευρώπη για τους πολίτες, να επαναφέρουμε σε αύξηση 10% τις σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού, τα σχετικά κονδύλια. Ένα ποσό το οποίο πιστεύουμε πως είναι αποδεκτό και για την Επιτροπή των Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου και που θα αποτελέσει το μήνυμα εκείνο που θα αποστείλουμε στο Συμβούλιο για να πούμε ότι δεν δεχόμαστε ε, περικοπές και επιπλέον θέλουμε ενίσχυση των κονδυλίων και έτσι μπορούμε να ξεκινήσουμε μια βάση διαπραγμάτευσης για τον τριμερή διάλογο. Στα πιλωτικά προγράμματα και τα υποπροετοιμασία μέτρα. Κάθε τροποποίηση στον προϋπολογισμό παρακαλώ να αφορούν μόνο εκείνα τα ε, έργα στα οποία η Επιτροπή έχει δώσει αξιολόγηση α ή β. Πράγμα το οποίο σημαίνει πως η Επιτροπή φρονεί πως ε, είναι δυνατόν να υλοποιηθούν είτε απευθεία τα α, είτε σχετικά εύκολα τα κατηγορία Β. Να μην ε, επιμείνουμε δηλαδή για προγράμματα στα οποία δεν έχουμε καμία ελπίδα επιτυχίας. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω τα προγράμματα α και β θα προτιμούσα να ε, είναι αυτά τα οποία θα υποστηρίξουμε. Βέβαια έχετε κάθε ελεύθερο εσείς να υποβάλλετε τις τροπολογίες που σας ενδιαφέρουν. Για, για τα προγράμματα τα οποία η Επιτροπή έχει χαρακτηρίσει με το Β, έχει εντάξει την κατηγορία Β, χρειάζεται μια επιπλέον αξιολόγηση και μετά μπορούμε να δούμε αν μπαίνουν στον προϋπολογισμό. Αλλά πάντως δεν ε, θα υποστηρίξω εγώ ε, προγράμματα ή έργα τα οποία η Επιτροπή έχει χαρακτηρίσει ως σε ΙΝΤΕ. Βέβαια αυτό θα το αποφασίσουμε συλλογικά στην Επιτροπή. Για τα πιλωτικά προγράμματα και τις πληροφορίες για αξιολόγηση που θα μπορούσαμε να δώσουμε στην Επιτροπή. Παρακαλώ να κοιτάξουμε τις ε, προτάσεις που θα κατατεθούν, να τις καταθέσουμε μέχρι τις 25 του μηνός και εφόσον προχωρήσει το χέτερο δυνατό η αξιολόγηση αυτή από την Επιτροπή, να έχουμε την ευκαιρία να εξετάσουμε αν τα διατηρούμε ή αν τα αποσύρουμε τα μέτρα αυτά ή τα έργα. Ιδάλλως δεν θα μπορέσουμε να τα εντάξουμε στο έτος. Δυστυχώς. Βεβαίως περιμένω τις περαιτέρω προτάσεις σας, τροπολογίες, ιδέες για τον προϋπολογισμό. Πάντως πιστεύω ή ελπίζω τουλάχιστον να γίνουν δεκτές οι δικές μου προτάσεις ε, και από εσάς. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και περιμένω τις, ε, τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κάμερεβερτ. Ε, θα ήθελα, προτείνω το εξή. Πρώτα απ' όλα να λάβουν το λόγο, θα έλεγα, οι σκιώδει ηγητέ. Αλλά ξέρετε κάτι, ο κύριο Κρίστιαν Έιλε, που είναι ο μόνος σκιοδησηγητής που είχε πει ότι θα τοποθετεί, δεν είναι παρόν. Και οι άλλε πολιτικέ ομάδε δεν έχουν ακόμα προτείνει ηγητή. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω του συντονιστέ να ορίσουν ηγητέ ε, το συντομότερο δυνατόν. Μέχρι τις 25 Ιουλίου έχουμε χρόνο ε, και οι συζητήσει θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τι αρχέ Σεπτεμβρίου για να ξέρουμε τι θα κάνουμε με το θέμα αυτό. Πρέπει εντωμεταξύ να έχουν ε, δρομολογηθεί και οι συμβιβασμοί, πρέπει να έχουν οπωσδήποτε οριστεί οι σκιώδει Παρακαλώ τι πολιτικέ ομάδε να τοποθετηθούν. Euh, Εμείς ορίσαμε σκιώδη εισηγήτρια στην ομάδα μου. Εμένα. Ωραία. Θέλετε να μιλήσετε κατευθείαν. Θα, ενημερώ, θα επικοινωνήσω και θα ενημερώσω σχετικά την κυρία Καμεραβέτ μέσα στη εβδομάδα. Άλλη για τον προπολογισμό, η κυρία Μπίλντε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βλέπω μια διασπορά πόρων ξανά. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπαίνει σε μια περίοδο Δημοσιονομική αβεβαιότητα λόγω του Brexit. Δεν είμαι ιδίω υπέρ της συνέχισης του προγράμματος Discover EU που, προβλέπει, που προτείνει ε, εισιτήρια τρένων για 18 χρονούς με μείωση 13 εκατομμυρίων ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών. μείωση 162 εκατομμύρια ευρώ για το Ευρωπαϊκό Σώμα Πολιτικής Ασφάλειας και Αλληλεγγύης δεν νομίζω ότι είναι, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά υπερβολικά. Η, τα ποσά που δίνουν για την εκτελεστική επιτροπή παραμένουν ε, χωρίς αλλαγή. Δεν πρέπει να διασπαθίζουμε τους λίγου πόρους της Ένωσης σε ε, μικρές και διαφοροποιημένες αποστολές εκτός και εντός της Ένωσης όπως συνέβη συχνά στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Κύριε Γιουρέκ. Ήθελα να πω ότι αύριο, μέχρι αύριο θα έχουμε αποφασίσει για το σκέο τη ηγητή. Εμείς μέχρι αύριο τα ξέρουμε. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω. Και δεύτερον, θέλω να πω ότι πρέπει πραγματικά να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα καλύτερο προϋπολογισμό για την Επιτροπή μας. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει με εμά, ο τρόπος που μας μεταχειρίζονται. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, θέλει κανείς άλλο το λόγο. Ντινόλφη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Σωστά τα λόγια του συναδέλφου. Είδαμε ότι τα προηγούμενα πέντε χρόνια οι πόροι της Επιτροπής μας ήταν πάντα πόροι για τη τακτομπούτα. Ποτέ δεν είχαν ε, ουσιαστική έμφαση. Αντίθετα, ο πολιτισμός ως εκπαίδευση, ως διδασκαλία των πολιτών, ως επίγνωση των πολιτών, είναι από τις μεγάλες υποχρεώσεις ε, της Ένωσης και πρέπει να παροτρύνουμε ούτω ώστε όλα τα προγράμματα της Επιτροπής Πολιτισμού, ιδίως το Creative Europe, ε, που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για τους πραγματικούς δημιουργούς και να δώσουμε μεγαλύτερη χρηματοδότηση από την Ένωση. Για τα πιλωτικά σχέδια, ξέρουμε ότι τα σχέδια που έχουν μια αξιολόγηση B, C και D πολλές φορές, σχεδόν πάντα, δεν χρηματοδοτούνται, δεν λαμβάνονται καν υπόψη. Αυτό είναι κρίμα, διότι μέσα στα πιλωτικά σχέδια μπορεί να υπάρχουν και ενδιαφέρουσες ιδέες που θα μπορούσαμε να προτείνουμε σε πολίτες και ενώσεις. Εμείς ως κίνημα πέντε αστέρων θα προτείνουμε εκ νέου το Media Literacy ως πιλωτικό σχέδιο, ένα πρόγραμμα που λειτουργήσε πολύ καλά στο παρελθόν και που δείχνει τη σημασία, είναι σημαντικό για να μπορέσει να προχωρήσει σε, ψηφιακή, σε ψηφιακό αλφαβητισμό για την καταπολέμηση του fake news και για την καλύτερη κατανόηση το πώς αυτά τα νέα τεχνολογικά μέτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα. Ευχαριστώ την Περβία και ελπίζω την επόμενη πενταετία να συνεργαστούμε με αποτελεσματικό και θετικό τρόπο. Η κυρία Σόντροβα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ εντάχει στο, στις επικρίσεις που ακούστηκαν για το Erasmus και το Creative Europe. Εμείς διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλοί δυσαρεστημένοι ακόμα. 20% μόνο πηγαίνει σε τέτοια σχέδια ε, το θέμα είναι να υπάρχει καλύτερη κινητικότητα των φοιτητών και των καθηγητών. Μιλάμε για δημιουργίες ε, πραγματικών πνευματικών δημιουργών που πηγαίνουν σε πραγματικά χρήσιμες δράσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, πρόκειται για μια πρόταση εξαιρετικά χρήσιμη και σημαντική γιατί λαμβάνει υπόψη το ότι υπάρχει μια εκδήλωση ενδιαφέροντας από πλευρά νέων και εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπάρξει μια ουσιαστική χρηματοδότηση. Ταυτόχρονα συμφωνώ και ότι είναι χρήσιμο για τον ε, αλφαβητισμό και την αύξηση της εγγραμματοσύνης. Ο Φραντς, για μένα είναι σημαντικό να έχουμε κατά και το παρελθόν, δηλαδή να γνωρίζουμε στο παρελθόν τι ακριβώς έγινε με την βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων. Η δική μου η εμπειρία είναι η εξή ότι πολλοί πολίτες στην Ευρώπη, πολλοί παραλαμβάνω, ε, δεν ήταν σε θέση να συμμετάσχουν σε προγράμματα, γιατί τα εμπόδια ήταν πάρα πολύ ψηλά Αλλά γνωρίζουμε ότι τα προγράμματα τα οποία ξεκινούν από πάνω, από την κορυφή και βαδίζουν προς τα κάτω, προς τη βάση, αυτά δεν είναι επιτυχημένα. Ως εκ τούτου, και αυτό έχει αποδειχθεί και από άλλες περιπτώσεις, ε, είναι καλύτερα, τα προγράμματα ξεκινούν από τη βάση προς τα πάνω αντιπατερναλιστικά προγράμματα, αυτά είναι τα καλά, αυτά λειτουργούν. Και γνωρίζετε ότι κατά παρελθόν είχαμε και την ε, έκθεση για τους Ρωμά, η έκθεση τελικά δεν ε, είχε μεγάλη αποτελεσματικότητα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί, τους οποίους αφορούσε η έκθεση, αυτοί δεν αντιμετωπιστήκαν ως ίσοι. Και αν πραγματικά θέλουμε βιωσιμότητα και θέλουμε να είμαστε ε, επιτυχημένοι και θέλουμε πραγματικά να αλλάξουμε την ε, θέση των ε, ανθρώπων που μενεκτούν σε επίπεδο πολιτισμού, τότε θα πρέπει να μειώσουμε τα εμπόδια, να αρχίσουμε να συμπεριλαμβάνουμε τους ανθρώπους που είναι οι άμεσα θυγόμενοι και με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά τη διαφθορά και να είμαστε και πιο επιτυχημένοι. Αυτό αποδεικνύουν τα προγράμματα τα οποία έχουμε εξετάσει. Αυτή είναι η εμπειρία μας. Και τώρα όσον αφορά τα πιλωτικά μας προγράμματα, πρέπει να σας πω, ότι τα διάβασα πολύ προσεκτικά και διαπιστώνει κανείς εκεί ότι όσοι αποφασίζουν δεν έχουν τις γνώσεις για το τι συμβαίνει επί τόπου και γι' αυτό ίσως να μην λαμβάνονται και οι σωστές αποφάσεις. Γι' αυτό λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι να μιλήσουμε ακριβώς γι' αυτό το πώς ε, μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε όσοι είναι αρμόδιοι στη διοίκηση για τη λήψη αποφάσεων, έτσι ώστε να λαμβάνονται οι σωστές αποφάσεις. Αυτό είναι εκείνο που εύχομαι κατά την επόμενη, την τρέχουσα θητεία, ότι θα τα καταφέρουμε όλοι από κοινού. Ο κύριος Βίνκλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πραγματικά είμαι ενθουσιασμένος που είμαι έστω και αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή αυτή. Ελπίζω η εντολή που ψηφίσαμε πριν από λίγο θα υλοποιηθούν σωστά από την ομάδα διαπραγμάτευσης και ότι θα έχουμε επαρκή κονδύλια τα επόμενα χρόνια και για το Εράσμους και συνολικότερα ταυτόχρονα να εκφράσω την ελπίδα μου ότι τα προγράμματα που απευθύνονται στους νέους θα χρηματοδοτηθούν πολύ καλά και να βρούμε συνέργειες μεταξύ των υφιστάμενων προγραμμάτων. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πραγματικά είμαι ενθουσιασμένος με αυτό το πρόγραμμα Bubble EU. Δεν είναι ένα τυχαίο μικρό, μικρό μικρή σημασία γεγονός. Είναι ένα δείγμα το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται για τους νέους, ε, δηλαδή ακόμα και το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρει πως γίνεσαι 18, ξέρει πως 18 χρονών είναι σημαντικό για τους νέους αυτούς ε, που προσπαθούν, που μπαίνουν στην ενήλικη ζωή. Η υποστήριξη των νέων από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ μεγάλη σημασία. Προφανώ μπορούμε να το συνδέσουμε μέσω συνεργειών και με άλλα προγράμματα, π.χ. το Εράσμους. Αλλά καθήκον μα είναι να δαπανίσουμε πολύ περισσότερα κονδύλια για τους νέους μας και για τα προγράμματα για τους νέους. Ό,τι και να κάνουμε στον τομέα της επικοινωνίας, της αντιμετώπισης των νέων προκλήσεων, των fake news, είναι πράγματα που χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε ως νέα φαινόμενα. Δεν τα είχαμε πριν από 15-20 χρόνια. Πρέπει τα νέα αυτά προβλήματα να τα αντιμετωπίσουμε μαζί με τους νέους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Βίγκλερ. Τώρα λοιπόν θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Κομισιόν, γιατί δεν βλέπω να ζητάει κανείς άλλο το λόγο, αλλά πριν δώσω το λόγο στην Κομισιόν θέλω και εγώ να πω κάτι. Ε, σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα, α, μισό λεπτό, ε, θα σας δώσω αμέσως το λόγο. Ε, κοιτάξτε, έχουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο εξολογήθηκε με C, όχι βέβαια από την Δικη Επιτροπή, αλλά από τη Γενική Διεύθυνση Προπολογισμού. Ω εκ τούτου, και εγώ έχω την παράκληση να δείτε πολύ προσεκτικά και τα προγράμματα C, γιατί δεν αξιολογήθηκαν σωστά. Υπάρχει, α πούμε, ένα πιλωτικό project ε, το οποίο ε, έχει συμπεριληφθεί και στα νέα προγράμματα, άρα δεν μπορεί να είναι και τόσο χάλια που να αξιολογείται με «σι». Ε, το να το θεωρούμε εμείς ότι είναι καλό και το προτείναμε για τα νέα προγράμματα, κάτι δεν πάει καλά. Ως εκ τούτου σας παρακαλώ να ρίξετε μία ματιά σε όλα τα προγράμματα. Ο κύριος Λούις Ντεβέζα έχει στήσει το λόγο και μετά θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία αναφορά στο θέμα των πιλωτικών σχεδίων, όπως και εσείς πριν από ένα λεπτό. Μια γενική παρατήρηση καταρχάς, η έμφαση της εκπροσώπου της ομάδας μας, κυρίας Καμερβέτη, είναι πολύ σωστή. Τα προγράμματα αυτά είναι καθοριστικά, εξαιρετικά σημαντικά και ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξύ των πολιτών της Ένωσης. Αυτό συμβαίνει προφανώς με το Erasmus Plus. Είναι απαράδεκτο λοιπόν το Συμβούλιο να εξετάζει ενδεχόμενα περικοπών. Είναι προγράμματα που πρέπει να χρηματοδοτηθούν με περισσότερα κονδύλια από ό,τι τώρα. Μεταξύ αυτών και διότι είναι γεγονό και αυτό πρέπει να το δούμε στο μέλλον, οι συνθήκες δεν παραχωρούν στην Ένωση σοβαρές αρμοδιότητες στον τομέα με τον οποίο ασχολείται η Επιτροπή μας Εκπαίδευση και Πολιτισμού. Έχουμε ωστόσο αυτά τα προγράμματα. Εφόσον λοιπόν δεν έχουμε γερές αρμοδιότητες, σας έχουμε γερή χρηματοδότηση που θα έχει σημασία, μια και η Ένωση μπορεί να προχωρήσει μόνο στην... δεν μπορεί να προχωρήσει μόνο με την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών ή... αλλά και με μεταρρύθμιση των συνθήκων που πρέπει να δούμε στη θητή αυτή. Ε, παράλληλα ωστόσο πρέπει να ενισχύσουμε την έννοια της ευρωπαϊκής ηθαγένειας πολιτιστικά και εκπαιδευτικά. Για τα πιλωτικά τώρα που σχολίασε και η Πρόεδρος. Υπάρχει κάποιο που η Επιτροπή συνεχίζει να χαρακτηρίζει ως σε, σε όλες τις περιπτώσεις που το υποβάλλουμε. Τρίτη τέταρτη περίπτωση, τρίτη φορά είναι. Δεν ξέρω αν θέλει να σχολιάσει αυτό η Επιτροπή. Μια πρόταση βοήθειας στην εφαρμογή ενός προγράμματος που εντοπίζει σε κάθε Δήμο της Ένωσης έναν σύμβουλο, ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου που θα είναι αρμόδιος για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων κατάρτισης και συζητήσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα είχε πολύ μεγάλη σημασία σε κάθε επίπεδο και θα έφερνε την Ευρώπη πιο κοντά στον πολίτη, στο Δήμο, στο επίπεδο του Δήμου και της κοινότητας. Γιατί λοιπόν η Κομισιόν έχει φαγωθεί να το χαρακτηρίζει ως σε τρεις-τέσσερις φορές, ενώ υπάρχουν προγράμματα που ήδη ασχολούνται με το θέμα αυτό και που δεν ε, αποδίδουν ε, σωστά. Ευχαριστώ. Η κυρία Γουόρτ. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να λάβω το λόγο για να υπερασπιστώ την επένδυση που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που κάνει ακόμα μέσω των προγραμμάτων για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση στις σχέσεις με τις τρίτες χώρες. Θα αναλάβετε όλοι σας αρμοδιότητες, θα λάβετε μέρος σε αντιπροσωπείες για σχέσεις με τρίτες χώρες και όταν ε, θα είστε μέλη τη αντιπροσωπή αυτέ, δεν πρέπει να λησμονείτε ότι είστε και μέλη τη Επιτροπή Πολιτισμού. Και όταν πηγαίνετε στι χώρε αυτέ, να του ρωτάτε, ρωτάτε τι κυβερνήσει και του αξιωματούχου για τα προγράμματά του για τον πολιτισμό και να δείτε ε, η διεισόμαση, την ε, εφαρμογή στην πράξη αυτών των συνεργατικών σχέσεων το λέω αυτό διότι είχα την ευκαιρία και μέσω της αντιπροσωπείας για τη Βοσνία Ζεγοβίνη και το Κοσμοπέδιο στην τελευταία θητεία να ε, διαπιστώσω τι συμβαίνει και ξέρω πόσο τεράστια αλλαγή μπορεί να επιφέρουν τα κονδύλια των, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση σε χώρες που έχουν βγει από εμπόλεμες καταστάσεις. Μιλείς μόνο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρώτα αρχικά και πάνω απ' όλα ε, ένα έργο ειρήνης και αυτό μπορούμε να προσφέρουμε στις χώρες αυτές μέσω του πολιτισμού, μέσω της προσέγγισης στην ανθρωπιά, στην, ε, στις παραδόσεις κτλ. Ε, να προσεγγίσουν ένα τον άλλον και γι' αυτό δεν υπάρχει ούτε ευρώ που πηγαίνει χαμένο από τα προγράμματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Judy Ward, κοιτάω να δω πώς θέλει κανείς το λόγο. Αν όχι, η Επιτροπή παρακαλώ για να τοποθετηθεί. Ποιος εκπροσωπεί την Επιτροπή σήμερα. Παρακαλώ. Το μικρόφωνο δεν λειτουργεί. Το μικρόφωνο δεν λειτουργεί καθόλου. Because it's not working. please switch off the... Uh, okay, thank you very much for... Σας ευχαριστώ πολύ και στο συγγνώμη για το λάθος μου το μικρόφωνο. Πιστεύω τώρα να δουλεύει. Ήθελα ξεκινώντα να συγχαρώ την Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους, αλλά και όλη την Επιτροπή Πολιτισμού και εκπαίδευση ε, για τη νέα θητεία και εύχομαι κάθε επιτυχία στα σημαντικό έργο σας. Επί τη ευκαιρία ευχαριστώ και την ε, απερχόμενη πρόεδρο, κυρία Καμερέβερτ, για την εξαιρετική δουλειά που έκανε ω πρόεδρο τη Επιτροπή τα τελευταία χρόνια, υποστηρίζοντα την πολιτική και τα προγράμματα τη γενική μα διεύθυνση, που είχαν πολύ μεγάλη σημασία για τι πολιτικέ μα και κρίσιμη. Για τον προπολογισμό του 2020, πρέπει να είμαστε βέβαιοι πω κάθε ευρώ του ευρωπαϊκού προπολογισμού εξασφαλίζει προσθέμενη αξία για τον Ευρωπαίο πολίτη. Αυτό είναι εκ κάνευ προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γενικότερα, αλλά και για την γενική μου διεύθυνση και το κεκτημένο επίσης ε, για την περίοδο 2027 πρέπει να εξασφαλιστεί. Ε, είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να υπολογίζουμε στην υποστήριξη της Επιτροπής σας και ε, ότι θα συνεχίσουμε την επικοδομητική και αποτελεσματική συνεργασία. Ο προπολογισμό αυτός, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο του 2020, είναι μάλλον το, ο προπολογισμό για το 2020 είναι ο τελευταίο τη επταετία που ξεκίνησε το 2014 και θα ε, έχουμε σαν προτεραιότητα την ανταγωνιστική οικονομία αλλά και τις ε, ε, δημιουργικές ε, δραστηριότητες με εστίαση στους νέους. Έχουμε ένα έτος δημοσιονομικό που έχει ξεκινήσει σε χαμηλά επίπεδα το 2014, αλλά παρουσιάζει μια γεωμετρική ανάπτυξη χρόνο το χρόνο. Έτσι το 2020 είναι κρίσιμο έτος για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την κάλυψη όσο δυνατόν περισσότερων προγραμμάτων, προγραμμάτων που μέχρι τώρα δεν είχαν χρηματοδοτηθεί σε τέτοιο όγκο στην περίοδο αυτή του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και να ανοίξουμε και άλλα θέματα. Και θα ήθελα και γι' αυτό να σας ευχαριστήσω για την εκκίνηση του διαλόγου από εδώ και μπρο. Έχουμε από την άλλη λοιπόν ένα πολύ σημαντικό θέμα για την προσεχή περίοδο. Από το 2020 ο προπολογισμό 2020 πρέπει να οριστεί ως το απόλυτος ελάχιστο ποσό που θα ε, προχωρήσει στο σχεδιασμό της επόμενης ε, δημοσιονομικής περίοδου. Γι' αυτό λοιπόν έχουν πολύ μεγάλη σημασία αυτά που λέγονται εδώ, να εξασφαλιστεί δηλαδή η συνεργασία που ανέκαθεν υπήρχε μεταξύ της Επιτροπής σας και της ε, υπηρεσίας της δικής μας ε, των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020 το πρόγραμμα Εράσμους ισχύει την ε, χρηματοδότηση των εταιρικών σχέσεων, της κινητικότητας στο τομέα της ανώτερης εκπαίδευσης, στην δευτεροβάθμια και γενικά στην νεολαία με 56 εκατομμύρια επιπλέον ευρώ για τον επόμενο προϋπολογισμό οι οι πιστώσεις θα είναι 1,63 συνολικά δισεκατομμύρια. Θα έχουμε επίσης το πρόγραμμα Erasmus Plus που θα επιτρέπει και δράσεις κοινωνικής συμπερίληψης διεθνικών και εθνικών δικτύων σε συνεργασία με υπηρεσίες παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης στους νέους και τους ενήλικες, ε, επαγγελματική και ε, διαρκή κατάρτιση και αριστεία στην κατάρτιση που άλλωστε έχει ζητήσει και η Επιτροπή σας. Το Δημιουργική Ευρώπη. Και θα πρέπει να αγωνιστούμε για να εξασφαλίσουμε καλά αποτελέσματα μετά το Συμβούλιο για να μην περικοπεί το πρόγραμμα. Καθώς έχουμε σχετικά μη ικανοποιητικά επίπεδα επιτυχίας τα τελευταία χρόνια. Πρέπει λοιπόν αυτές οι οργανώσεις να ενσωματωθούν για να εξασφαλιστεί το απαραίτητο επίπεδο χρηματοδότηση που όπως είπα δεν ήταν ικανοποιητικό. Η γραμμή αυτή του προϋπολογισμού, Δημιουργική Ευρώπη, επιτρέπει τη συνεργασία πάνω από 100 διαφορετικών οργανώσεων ανά την Ευρώπη, μικρές και μεσές οργανώσεις συνολικά. Και αυτή είναι η επισκόπηση του Σχεδίου προπολογισμού 2020, τομείς προτεραιότητας που εξετάζουμε για τα κύρια προγράμματα, το Erasmus Plus, το Σώμα Αλληλεγγύης και τη Δημιουργική Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, και θα ήθελα σε αυτή τη ε, σε αυτό σημείο να σημειώσω ότι ό,τι ακούσατε, ό,τι συζητήσαμε εντάσσονται ακριβώ στο πλαίσιο των όσων έχουμε μέχρι τώρα συμφωνήσει στο τελευταίο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Ξεκινούμε δηλαδή με το, η πρώτη χρονιά με χαμηλότερη χρηματοδότηση, έτσι ώστε να ξεκινήσουν τα προγράμματα και να ολοκληρωθούν τα προηγούμενα. Και άρα ό,τι έχουμε προτείνει καλυπτόταν τους άλλους από το πρόγραμμα. Κυρία Κάμερα, ευχαριστώ πολύ. Πολύ σημαντική επισήμανση αυτή σε όλα τα προγράμματα. Ξεκινήσαμε με λιγότερα χρήματα γιατί έπρεπε ούτως ή άλλως ή μπορούσαν μάλλον να τεθούν σε πλήρη λειτουργία τα προγράμματα αργότερα γιατί είχαμε και την εκκρεμότητα με το πολιτισμο νοσονομικό πλαίσιο και έτσι οι αυξήσεις είδαμε ότι ήρθαν σύν το χρόνο, χωρίς να σημαίνει όμως ότι πήραμε επιπλέον ποσά από είχαν αρχικά προϋπολογιστεί. Τώρα, οι περικοπές που το Συμβούλιο και για το Δημιουργική Ευρώπη και για το Μέντια και για τον πολιτισμό αλλά και για το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες ε, είναι τελείως απαράδεκτες αυτές οι περικοπές του Συμβουλίου. Τα 6 εκατομμύρια που θα μπορούσε να εξοικονομήσει συνολικά στον προπολογισμό δεν έχουν κανένα αντίκτυπο, ελάχιστο αντίκτυπο, ε, ενώ επιφέρουν ε, βαρύτατο πλήγμα ακριβώς εκεί όπου προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε την συμμετοχή του πολίτη, την υποστήριξη του πολίτη για την Ευρώπη, εκεί όπου μικρές και μεσαίες, μεσαίου μεγέθους πρωτοβουλίες και έργα για τον πολιτισμό ή οπτικοακουστικά προγράμματα ε, και δραστηριότητες στην Ευρώπη θα μπορούσαν να ενισχυθούν. Λυπούμε πολύ γι' αυτό είναι προφανέ ότι, τουλάχιστον έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ την κατάσταση, η πλειοψηφία των συναδέλφων εδώ στο Κοινοβούλιο ε, αντιτίθεται σε αυτή την πρόθεση του Κοινοβουλίου και με ακολουθεί στην πρόταση για ε, διεκδίκηση μιας αύξηση 10% των ε, ε, ποσών για όλα τα προγράμματα αυτά, έτσι ώστε να έχουμε καλές ε, πιθανότητες επιτυχίας και να δώσουμε και το κατάλληλο μήνυμα για τα πιλωτικά προγράμματα. Βεβαίως υπάρχουν καλές ιδέες, ευφύης ιδέες στα πιλωτικά προγράμματα, το ξέρουμε πολύ καλά αυτό, ταυτόχρονα όμως ξέρουμε ότι είναι ε, περιορισμένα τα μέσα που είναι διαθέσιμα για τέτοιου είδου πιλωτικά έργα. Είμαι διατεθειμένη βεβαίως πάντα να κοιτάξω για άλλη μια φορά εάν υπάρχει δυνατότητα σε κάποιο έργο που ενδεχομένως να αξιολογήθηκε με τρόπο εσφαλμένο να γίνει κάποια διόρθωση. Πάντως για μας οι προτεραιότητες πρέπει να προσδιοριστούν αμέσως γιατί αν δεν τις ορίσουμε εμείς τις προτεραιότητες θα τις ορίσουν κάποιοι άλλοι και δεν θα είναι αυτές που θέλουμε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να έχουμε βρει και μια σωστή και λογική γραμμή. Για τι συνομιλίε. θα αγωνιστούμε θα παλέψουμε σκληρά. Στον τριμερή διάλογο θα επιδιώξουμε διπλασιασμό των μέσων όπω έχει στήσει το Κοινοβούλιο τη Δημιουργική Ευρώπη και τριπλασιασμό των κονδυλίων για το Erasmus Plus και διπλασιασμό του προγράμματο για το Ευρώπη των πολιτών. Ε, θα είναι σκληρό ο αγώνα, σκληρή η μάχη το ξέρουμε. Ωστόσο, το Κοινοβούλιο παγίως επισημαίνει ότι η μεγάλη αξία που αποδίδει στο να είναι για τον ετούντα απλές οι διαδικασίες στην διαδικασία της κατάθεσης ε, μιας ε, αίτησης για συμμετοχή σε προγράμματα, γιατί πάντα αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και εμείς επισημαίνουμε ότι συχνά οι πολίτες οι ενδιαφερόμενοι βλέπουν με δυσφορία ότι δεν, δεν δίνεται υποστήριξη στα μικρά προγράμματα όπως θα ήθελαν. Δεν τους ενδιαφέρουν δηλαδή τα μεγαλεπίβολα έργα πολιτισμού, αλλά τα πιο μικρά, τα πιο στιγμιαία ε, πολιτιστικά έργα. Αυτά τα οποία ακριβώς μπορεί να επιτρέψει το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη να ε, δουν το φως. Περιμένω βέβαια τις προτάσεις ε, του Συμβουλίου για να τις αξιολογήσω και είμαι βέβαιη ότι θα χρειαστεί και να τις ε, αποκρούσω. Ε, πιστεύω ότι εμείς εδώ απαιτείται να αναλάβουμε δράση. Είναι απαραίτητο να έχουμε περισσότερα κονδύλια για τους τομείς δραστηριότητας της Επιτροπής μας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ την ε, κυρία Πέτρα Κάμερεβερτ. Ε, δεν βλέπω να θέλει κάποιος άλλος το λόγο. και κανονικά και μετά την εισηγήτρια κλείνει η συζήτηση. Ως εκ τούτου τελειώνουμε τη συνεδρίασή μας. Ε, το μόνο που μου απομένει είναι να σας επαναλάβω την 25η Ιουλίου, 4 ώρα το απόγευμα, καταληκτική ημερομηνία για κατάθεση τροπολογιών. Παρακαλώ στα αγγλικά. Η επόμενη συνεδρίαση, Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου, 9 με 6.30 και την 5η 5 Σεπτεμβρίου 9 με 12.30. Το μόνο που μου απομένει είναι να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές και να μας επανέλθετε στις Βρυξέλλες υγιείς και χαρούμενοι. Τα λέμε το Σεπτέμβριο. Γεια σας. Και ευχαριστώ και πάλι τους και τις διερμηνείς και καλές διακοπές εύχεται η Πρόεδρος τους διερμηνείς.